Κυρία Γκρέσλε, είστε έτοιμοι? You have to knock. collègues, Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Κυρία Γκρέσλι είναι έτοιμη για την αναβολή. Madame Έχετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε, για τους νέους ε, κανόνες ε, που ισχύουν για το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Με συγχωρείτε, αλλά με πιάσατε εξαπίνης. Δεν ήξερα ότι είναι η σειρά μου ότι έφτασε όλας. Μάλιστα, θα συνεχίσω στα γερμανικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον ε, προϋπολογισμό. Εγώ κατόρθωσα να ολοκληρώσω την έκθεση, κάπως καθυστερημένα τώρα, είναι υπομετάφραση. Βέβαια έχει διανεμηθεί το αγγλικό κείμενο, 18 Ιανουαρίου και θα έχουμε μία συζήτηση στις 20 Ιανουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και κατόπιν θα έχουμε και τις τριμερείς συναντήσεις, θα έχουμε και δύο γνωμοδοτήσεις από τις Επιτροπές Σέντε και ΑΦΕΤ και επίσης ο συνάδελφος Ντάμας Ντόιτς επίσης ε, θα καταθέσει μια γνωμοδότηση και κάποιος άλλος συνάδελφος. Έχω μιλήσει με δύο εισηγητές και έχω υιοθετήσει όσα μπορώ. Επίσης, ε, συναντήθηκα με την ομάδα εργασίας ε, για να συζητήσουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και είχαμε συναντήσεις ε, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όταν θα καταλήξουμε σε συμβαστικό κείμενο με το Συμβούλιο θα συνεχίσει η ομάδα εργασίας με τις συνεδριάσεις της. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί σε σχέση με τις ε, οδηγίες που αφορούν και τις δημόσιες προμήθειες. Τα κράτη-μέλη έχουν δύο χρόνια για να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την νομοθεσία αυτή. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ νέα νομοθεσία μέχρι το 2016. δημόσιες προμήθειες είναι στο επίκεντρο του θέματος. Η Κομισιόν έχει προτείνει να ε, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, να υπάρχουν ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, παραδείγματο χάρη να μπορούν να διορθωθούν και οι συμβάσεις αναδρομικά. Όλα αυτά θα τα δει και η Διαχειριστική Επιτροπή των Προϋπολογισμών, αλλά μπορούν να υπάρχουν ε, και τροποποιήσεις αν χρειαστεί. Τώρα, η Κομισιόν θέλει να διευρύνει τη βάση δεδομένων της, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρώμικου κρίματος, τις απάτες, διάφορες παρατυπίες. Όλες αυτές οι παρατυπίες θα πρέπει να υπάρχουν και να αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων. Υπάρχει όποιο ανησυχεί για το πώ χρησιμοποιούνται τα κονδύλια θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων και φυσικά όσοι έχουν κάνει απάτε στο παρελθόν δεν θα μπορούν να το πράξουν και στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ιδέα αλλά είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία. Υπάρχει δουλειά που γίνεται εδώ και 8 χρόνια για αυτή τη βάση δεδομένων και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Εγώ έχω κάποιες τροπολογίες ε, υποβάλει και θα ήθελα τώρα να σας τις παρουσιάσω. Ελπίζω ότι αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη αναθεώρηση αυτής της νομοθετικής πρότασης και να είναι και τελευταία ευκαιρία για μένα να υποβάλω τροπολογίες στην πρόταση. Έχω λοιπόν υποβάλει κάποιες τροπολογίες που ξεπερνούν αυτά που έχει προτείνει η Κομισιόν η τροπολογία μου υπαριθμών 2 έχει να κάνει με τη δυνατότητα να αναγνωριστούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεθνεί οργανισμοί. Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει μέσω αποφάσεως της Κομισιόν, αλλά τώρα αυτό πρέπει να γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξης και αυτό το κάνουμε για να μην έχουμε άνηση μεταχείριση των διάφορων οργανώσεων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, αν κάποιος έχει ταξινομηθεί ως διεθνής οργανισμός μπορεί να λάβει κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να περάσει από διαδικασία ε, δημοσίων ε, συμβάσεων. Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε λοιπόν ότι ένας διεθνής οργανισμός, αν θεωρείται τέτοιος, θα πρέπει να σέβεται για κάποια κριτήρια και φυσικά αυτά τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι η απλούστευση. Τώρα για την τροπολογία 23. Άρθρο 209 και τα αποτελέσματα της τελευταίας τρογγυλής τράπεζας της 30 Νοεμβρίου. Εδώ πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία. Ελπίζω όμως ε, να μπορούν όλοι να συμφωνήσουν με το συμβασμό. επόμενη τροπολογία αφορά την εσωτερική υπηρεσία της Κομισιόν για τους ελέγχους, για τους λογιστικούς ελέγχους. Η τροπολογία 11, συγκρούσεις συμφερόντων, άρθρο 107. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τις συγκρούσεις συμφερόντων ως ε, λόγο για να μπλοκάρονται κάποιοι από τη συμμετοχή στη διαδικασία. Η Transparency International μας ζήτησε να το συμπεριλάβουμε. Τροπολογία 13. Έχουμε εδώ μια αναφορά στο να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων των εταιριών, αλλά δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για λόγους προστασίας των δεδομένων. Αυτά τα προστατευόμενα δεδομένα επίσης θα πρέπει να διατίθενται και σε εμά. Τροπολογία 14. να έχουμε ε, την περίπτωση μπλοκή σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, διαφθοράς κτλ. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να μπλοκαριστεί ένας υποψήφιος από να λάβει ε, συμμετοχή στη διαδικασία για πέντε χρόνια ή ίσως και για πάντα. Έτσι λοιπόν κάποιος ε, μπορεί να μπει μόνιμα στο μαύρο κατάλογο στη χειρότερη περίπτωση. Η επόμενη τροπολογία αφορά τις ε, κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους ε, δεν συνεργάζονται στα πλαίσια της βάσης δεδομένων και αν υπάρχουν ζημίες που προκαλούνται στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι για να υπάρχει συνεργασία πρέπει να έχουμε και το μαστίγιο και το καρότο. Επομένως, ε, υπάρχει και μια ακόμη τροπολογία, τροπολογία 23, που αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τις ειδικέ εκθέσεις. Εδώ έχουμε ε, προτείνει μια επιταχυνόμενη διαδικασία και μια υποχρέωση για την Κομισιόν να λαμβάνει υπόψη όλα τα προβλήματα του ελεκτικού συνεδρίου, με συγχωρείτε όχι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όλα τα προβλήματα που επισημαίνει το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή την τροπολογία θα πρέπει να την εξετάσω εκ νέου, εγώ έχω υποσχεθεί να μιλήσω με τον επικεφαλής ελεγκτή, να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα και να βρούμε μια λύση. Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ε, την προθεσμία που έχουμε τώρα, δηλαδή από ε, την ε, κατάρτιση μιας έκθεσης μέχρι τη δημοσίευσή της. Έτσι λοιπόν η τροπολογία 23 δεν είναι έτοιμη ακόμη, θα την επαναδιατυπώσω, δεν είχα χρόνο να συζητήσω ακόμη με όλους όσους ήθελα να συζητήσω κατόπιν μηχανισμός αποκλεισμού που προβλέπεται από την Κομισιόν ε, στις της πράξης. Νομίζω ότι αυτές είναι ουσιαστικές τροπολογίες. 6, 8, 15 και 16. Το Συμβούλιο συμφώνησε μαζί μου εδώ και επομένω συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτή την οδηγία παρά να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύση. Υπάρχουν και άλλε τροπολογίες με τις οποίες έχω προσπαθήσει να κάνω πιο διαφανές το κείμενο ή να είναι πιο συμβατό με τα άλλα νομοθετικά κείμενα γιατί η τελευταία πρώτη Κομισιόν δεν είναι ιδιαίτερα καινούρια. Θα σα διαβάσω τώρα κάτι Πρόκειται για την τροπολογία 1, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 20. Όλες αυτές είναι τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες. Επομένως, Πρόεδρε, αυτά πάνω κάτω από μένα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν ε, και άλλες τροπολογίες από μένα γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να συστήσουμε αυτή τη βάση δεδομένων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχω υιοθετήσει τις προτάσεις ε, της Transparency International, αλλά επίσης έχω συνομιλήσει και με νομικούς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ζήτησα την άποψή τους, την γνωμοδότησή τους και περιμένω την απάντησή τους. Επίσης είμαι ε, ε μάλλον ευχαρίστως ε, να σας δώσω και άλλα στοιχεία αν το χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μας διευκρινίσατε ποιες είναι οι πιθανές βελτιώσεις αυτού του σχεδίου οδηγίας για να διευκρινιστούν οι δημόσιες συμβάσεις και να εξασφαλίζεται διαφάνεια. Άλλωστε μπορεί να συμβεί να μην γίνονται δεκτές οι προσφορές που παρουσιάζονται από τις επιχειρήσεις που δεν είναι ενήμερες στις πληρωμές τους, διότι δεν πρέπει να υπάρχει αθέμετος ανταγωνισμός. Αλλά για να μπορεί να επιβάλλει αυτές τις αρχές η Ευρώπη, πρέπει και η Ευρώπη να είναι ενήμερη στις πληρωμές της. Ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο για την έκθεση που μας παρουσίασε μόλις τώρα. Μας είπε ότι οι προθεσμίες για τις τροπολογίες είναι η 8η Ιανουαρίου και ότι στις 20 Ιανουαρίου θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και ότι στις 5 Φεβρουαρίου η Επιτροπή μας θα κληθεί να ψηφίσει για τις τροπολογίες και για το τροποποιηθέν κείμενο. Κανένας δεν ζητάει το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν, όχι, παρακαλώ το λόγο, έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμανικά. Η έκθεση έχει συνταχθεί πολύ καλά και υπάρχουν ορισμένε πτυχές τι οποίες θα ήθελα προσωπικά να υπογραμμίσω ε, στην τελική διατύπωση. Η διαφάνεια πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο στις τροπολογίες μας ε, τι είναι η διαφάνεια. Δεύτερον, οι κυρώσεις γίνεται λόγος για τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν από όσους δεν σέβονται τους ισχύοντες κανόνες. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις, ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εφαρμοστούν. Τα πράγματα δεν είναι αρκετά σαφή. Και αν κατορθώσουμε να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, αυτό θα είναι πολύ θετικό. Μιλάμε για ε, ε, μια μέγιστη χρονική περίοδο 5 ετών για να εφαρμοστούν αυτές οι κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις και ποια είναι η διάρκεια για άλλες κυρώσεις και πώς μπορεί να επιτραπεί ή όχι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, μιλήσαμε για εξωτερικό έλεγχο. Πώς μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα πότε χρειάζεται εσωτερικός έλεγχος και πότε πρέπει να γίνεται εξωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που μπορούμε να συντάξουμε μαζί. Η ιδέα είναι να γίνεται έλεγχος επί των δημοσίων οικονομικών και νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να βελτιώσει πολύ σημαντικά τον έλεγχο αυτό. Εμείς θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να συντάξουμε μια τέτοια τροπολογία και κατόπιν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε στους φορολογούμενους πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματά του, πώς δαπανήθηκαν τα χρήματά του και πώς έγινε σεβαστή νομοθεσία. Μια άλλη ιδέα, η Τράπεζα Δεδομένων, θαυμάσια ιδέα. Καλό είναι να γίνει αυτή η τράπεζα και γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτό το μέτρο. Αλλά από δική μας πλευράς θα πρέπει να δούμε πώς εκείνοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Δεδομένων συμπεριλαμβάνονται με βάση σωστά κριτήρια. Διότι δεν πρέπει να βρεθούμε μπροστά σε καταστάσει όπου εκείνοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην τράπεζα δεδομένων θα μπορούν να προσβάλλουν την απόφαση λέγοντα ότι ορισμένα κριτήρια δεν έγιναν σεβαστά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η διαδικασία να είναι σαφή. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ, κύριο Σαγκαγιέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά την προηγούμενη θητεία είχα την ε, χαρά να είμαι σκιώδη ηγητής των σοσιαλιστών και εργάστηκα μαζί με την κυρία Κρέσλε για τον κανονισμό του προϋπολογισμού και βήμα προς βήμα πλάτη με πλάτη αν θέλετε ε, διαπραγματευθήκαμε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που ελέγχθησαν και έχω επιφυλάξει ε, ε, σε ένα μόνο θέμα στον τροπολογισμό υπερθμών 22. Να πω το εξή. Αυτή η ρήτρα γενικής εξουσιοδότησης για τον περιορισμό δυνατοτήτων απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί έχω επιφυλάξει δεν συμφωνώ, διότι κατά τα τελευταία πέντε έτη ακούσαμε ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, οι οποίες εκθέσεις ε, θα τις χαρακτήριζα χωρίς κάποια κριτική, όχι με την έννοια ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, εξέταζε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με το Γάντι. Εγώ θέλω να πω το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, είμαστε πολιτικό όργανο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν όλα αυτά που προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο τα θεωρούμε θέσφατα και θέλουμε να ερμηνεύσουμε όλα τα άλλα απλά και μόνο για να ασκήσουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε περιορίζουμε μόνοι μας τη δυνατότητα πολιτικής τοποθέτησης. Βεβαίως στο ελεγκτικό συνέδριο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ε, προβλήματα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο αρχής. Εγώ όμως ε, ως ε, εκλεγμένος βουλευτής θέλω να μπορώ να σκώ κριτική, όπως το του χάρη άμεση βοήθεια για αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες στο θέμα αυτό, θέλω όμως να πω ότι επ' αυτού είμαι κάθετα διαφορετικής άποψης από ό,τι υπήρξε κατά το παρελθόν το ελεγκτικό συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ε, δεν, ε, δεν εκφράζει επιχειρήματα λογιστικής φύσεως, αλλά πολιτικά. Και εγώ ε, θεωρώ ότι όσοι διαβάζουν τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει να μπορούν να αξιολογούν πολιτικά την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν λοιπόν περιορίσουμε αυτό το δικαίωμα, τότε τις ειδικέ εκθέσεις ε, θα τις ε, περιορίσουμε σε εκθέσεις στις οποίες θα μπορεί να ασκηθεί καθαρά λογιστική κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της αφαιρούμε το δικαίωμα να τοποθετείται πολιτικά. Αυτό δεν το βρίσκω σωστό. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τοποθετείται πολιτικά. Εμείς είμαστε πολιτικό όργανο και είμαστε σε θέση να κρίνουμε κατά πόσον προβάλλεται ένα πολιτικής φύσεως επιχείρημα της Επιτροπής ή όχι. Ε, γι' αυτό υπάρχουμε εξάλλου και γι' αυτό αρκετά όριμοι είμαστε για να μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε αυτό το συγκεκριμένο ε, επιχείρημα της Επιτροπής ε, ε, δεν το εγκρίνουμε. Αλλά δεν θέλουμε να μεταθέσουμε όλο το βάρος υπέρ του ελεγκτικού συνεδρίου, όχι κάθε άλλο. Ε, γιατί υπάρχουν πολλοί που ισχύονται ότι με τον τρόπο αυτό θα αφαιρέσουμε πολιτικά δικαιώματα ή πολιτικές τοποθετήσεις και ως εκ τούτου εγώ δεν θέλω να είμαι αναγκασμένος να δέχομαι συλλήπτην όλες τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και να μην ε, μπορώ ε, να τοποθετούμε πολιτικά όπως η Επιτροπή. Κυρία Γκρέσλε, θέλετε να απαντήσετε στους δύο μιλητές, γνωρίζοντας ότι όπως και έχουμε προθεσμία μέχρι τις 8 Ιανουαρίου για να ολοκληρώσουμε τις τροπολογίες και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα στις 20 Ιανουαρίου, καθώς όπως σας είπα θα ψηφίσουμε στις 5 ε, Φεβρουαρίου. Θα είμαι πολύ σύντομη. Για τη βάση δεδομένων. Είπατε ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις στην περίπτωση αποκλεισμού από την Τράπεζα Δεδομένων. Όμως, ε, Υπάρχουν ποινικέ διώξει όταν το κράτο μέλο δεχτεί κατηγορίε για ξέπλυμα χρήματο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσει όμως, ε, εφόσον πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια, αυτή είναι η μόνη κύρωση που προβλέπουμε. Και αυτός ο αποκλεισμό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτή λοιπόν η Τράπεζα Δεδομένων αναγκάζει τα κράτη-μέλη σε περίπτωση ε, δημόσιων έργων ε, να υπάρχει Τράπεζα Δεδομένων. Και όσοι κράτη-μέλη μας εξαπατούν να εμφανίζονται σε αυτή την Τράπεζα Δεδομένων. Μέχρι τώρα εκεί εμφανίζεται μόνο μία εταιρεία, γιατί ξέρετε πράγματι το διαδικαστικό όλο αυτό, η διαδικασία αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίπλοκη, τι λειτουργεί τελικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με την Τράπεζα Δεδομένων και θέλω να ελπίζω ότι αυτό που έχει κατατεθεί λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα. Εμείς ως Κοινοβούλιο το 2006 υπό τη Φιλανδική Προεδρία κατά τη μεταρρύθμιση επιβάλαμε την Τράπεζα Δεδομένων και Βεβαίως αυτό ήταν κάτι που ποτέ δεν το ήθελε το Συμβούλιο και δεν λειτουργήσε και ποτέ. Εν τω μεταξύ όμως έχουμε κράτη-μέλη που μας στηρίζουν περισσότερο, άρα δηλαδή μπορούμε να το ξαναδρομολογήσουμε το θέμα. Πάντως δεν πρόκειται για κάτι το αμεληταίο, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτό ε, που είπατε πραγματικά είναι το πρόβλημα οι αποφάσεις ε, του δικαστηρίου τώρα. Σχετικά με την τροπολογία 22 για το ελεγκτικό συνέδριο. Κοιτάξτε, το δικό μας το πρόβλημα είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο βαθμολογήθηκε πολύ αρνητικά από ε, άλλους, από ομολόγους, διότι το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει και γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει αυτός που ελέγχει σε σχέση με τον ελεγχόμενο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ελεγκτικό συνέδριο δεσμεύεται μέχρι και τη δημοσίευση της άποψης επιτροπής. Δηλαδή αυτό που εμείς ε, ε, έχουμε κατά νου και συζητήσαμε. Βεβαίως και το ελεγκτικό συνέδριο ενδιαφέρεται πάρα πολύ να διαβουλεύεται με την επιτροπή και να ε, έρχεται ε, σε περίπτωση διαφωνίας σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους ε, θεσμούς. Ε, θα υπάρξει λοιπόν μια διαδικασία σε περίπτωση διαφωνίας. Τώρα όμως αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Δυόμιση μήνες χρειάζεται η Επιτροπή και αυτό είναι το πρόβλημα. Λέμε λοιπόν ότι κοιτάξτε, έχετε χρόνο δυόμιση μήνες και εφόσον απαντήσετε θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το ελεγκτικό συνέδριο μετά από δυόμιση μήνες πρέπει πρέπει να ε, δημοσιοποιήσει το ε, αίτημα. Εγώ δεν λέω ότι η συμπερίληψη κομισιών σε διαφωνίες ε, θα πρέπει να προβλέπεται για να χρονοτριβούμε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια ειδική έκθεση που αφορά σε μια έρευνα των προγραμμάτων αγροτικών περιοχών γιατί εκεί τα ποσοστά σφάλματος είναι τόσο υψηλά. Επειδή λοιπόν η Κομισιόν δεν το επιθυμεί αυτό, χρονοτριβεί κόλληση εργή. Και ακριβώς αυτό το θέμα εγώ λέω δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ικανοποιήσουμε και τις δύο πλευρές. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχουν όλοι τα ίδια όπλα. Το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό ενδιαφέρεται ακριβώς για το ίδιο. Πράγματι μπορούμε να περιορίσουμε το χρόνο Δηλαδή και για το ελεγκτικό συνέδριο να πούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί στο χρόνο. Εμείς ως νομοθέτες ε, καταθέτουμε με λεπτομέρειες ε, το νομοθετικό στοιχείο και η ε, σύγκριση ομολόγων καταλήγει στο εξή. Γιατί ελεγκτικό συνέδριο το επιτρέπεται αυτό. Όλοι θέλουμε να είναι ίσα τα όργανα. Και αυτό σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν οι Κομισιόν και το Λεκτικό Συνέδριο. Εγώ λοιπόν δεν φοβάμαι ότι θα υπάρξουν ε, συμπεράσματα που δεν τα επιθυμεί κανείς, όμως νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, το ελεγκτικό συνέδριο στη σχέση του απέναντι στους ελεγχόμουνες. Και πρέπει να σας πω ότι το έχω εξετάσει λιγάκι το θέμα, το τι θα γίνει ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί και το ελεγκτικό συνέδριο ήλπιζε να αποκομίσει πολλά περισσότερα. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο δικός μας ο ρόλος είναι να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του ελεγκτικού συνεδρίου και στην περίπτωση αυτή ε, θα πρέπει να παρατηθούμε από τη διαδικασία που προβλέπει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Χαίρομαι λοιπόν για τις ε, τροπολογίες. Αν κάποιος ε, έχει ερωτήσεις, να έρθει να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Très bien. et eh bien, voilà une invitation qui a été Je pense qu'on peut Πολύ καλά, το ακούσαμε αυτό, μια πρόσκληση που ακούσαμε. Μπορούμε να μείνουμε εκεί όσον αφορά το σχέδιο τροποποίηση του οικονομικού κανονισμού. Το λόγο έχει κύριο Σταρό για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης σχετικά με το, τα αλλιευτικά δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, πρέπει να οριστικοποιήσουμε τις ε, ε, συμφωνίες αλλίες με τη Δημοκρατία της Σενεγάλης, η καλή είδηση είναι ότι από πλευρά προπολογισμού οι πληρωμέ και οι δεσμεύσει είναι ίσε. Συνεπώ δεν έχουμε επιπλέον προβλήματα πληρωμών, αλλά τα χρήματα δεν είναι πολλά, είναι 9,61 εκατομμύρια. Η συμφωνία αναφέρεται ε, στην, στους τόνους για τον τόνο 14.000 τόνους ετησίως και το άλλο είναι ο μαύρος μερλούκος 2.000 τόνους το χρόνο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτά τοποθετούνται στα όρια ε, των πλεονασμάτων που υπάρχουν, δηλαδή τα χρήματα, ε, τα, τα που μπορούν να λιευθούν χωρίς να διακινδυνεύσουμε ε, τα αποθέματα ή μπορούν τα νέα πλοία να αλλιεύουν, αλλά μέσα στα όρια που έχουν προβλεφθεί. Τώρα, οι επιστημονικές συμβουλές είναι κάπως, κάπως αντιφατικές όσον αφορά τον Μερλούκο. Και δεν υπάρχουν πολλά αποθέματα που να μπορεί να αλλιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαχείριση του, του Μερλούκιου θα πρέπει να γίνεται ε, με περιφερειακή βάση. Αυτό όμως είναι προβληματικό ε, σκέλος της συμφωνίας. Και δεν νομίζω ότι από τεχνική άποψη θα πρέπει η δική μας Επιτροπή να ασχολείται, αλλά μάλλον η Επιτροπή Ελίας. Συνιστώ λοιπόν η Επιτροπή Προπολογισμού να εκτιμήσει θετικά τη συμφωνία, διότι δεν νομίζω είναι θέμα χρηματικό θα ήθελα να σας δώσω κάποια τροφή για σκέψη, ορισμένες ιδέες που μπορούμε να περιλάβουμε στην γνωμοδότηση, διότι ε, είναι πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε να κάνουμε μια αλληλευτικές συμφωνίες υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη κυρώσεων όταν τα σκάφη δεν σέβονται ε, τις ζώνες αλίας. Πρέπει να να φροντίσουμε να σέβονται τα όρια που προβλέπονται ε, στους κανονισμούς. Όταν δεν συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσει, δεν θα πρέπει να τους δίνονται άδειες αλίας για τα σκάφη των κρατών μελών που δεν σέβονται τις συμφωνίες. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι η γραμμή προπολογισμού που αφορά την ληφτική Συμφωνία έχει υπερδιπλασιαστεί ε, διότι υπάρχουν ορισμένε μεταφορές. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των αλληλευτικών δραστηριοτήτων των χωρών γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναμενόταν. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί προβλήματα ε, διότι ε, γιατί θα υπάρχουν πλεονάσματα, δεν υπάρχουν πλεονάσματα ευθείων. Γι' αυτό θα πρέπει να... Τα όσα συμβαίνουν δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά ελιεύματα. Ε, τα οποία είναι ε, υπερδιπλάσια από την, χωρι... την χωρητικότητα αναφορά. αυτά είναι θέματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για το μέλλον και δεν θα πρέπει να μας εμποδίσουν στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Από ό,τι κατάλαβα, η προθεσμία για την, καταβολή ε, την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 18η Δεκεμβρίου και η συζήτηση μπορεί να γίνει στις 19 Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 9 Δεκεμβρίου και η οφέτηση θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας. Τώρα για την έκθεση του κυρίου Ταρά έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Τότε θα ζητήσω τον κύριο Γκάιερ αν θέλει να μας παρουσιάσει την εκθεσή, του για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία της ΕΠΟΛ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ευχαριστώ να σας μιλήσω για τη ΕΠΟΛ. Κοιτάξτε, εγώ έχω σπουδάσει ιστορία. Και αν δω λιγάκι τη μοίρα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών ε, μου έρχονται κατά νου ε, τα νόθα παιδιά του Μεσαίωνα που υπήρχαν αυτά και κανείς δεν τα ήθελε. Ήταν επιθύμητα. Σε προλ, λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία, Αστυνομική Ακαδημία που υπάρχει για την περαιτέρω κατάρτιση ε, των αστυνομικών αρχών των 28 κρατών μελών. Έτσι ώστε σε περίπτωση ε, διασυνοριακών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του εγκλήματος να είναι πιο αποτελεσματική. Τραγική η ιστορία αυτής της Ακαδημίας. Μετά από πολλά χρόνια που ήταν ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο ΣΕΠΟΛ ε, μετατέθηκε και Κατά την τελευταία θητεία συζητήσαμε σε βάθος για το θέμα αυτό. Ήταν μια συζήτηση που αφορούσε περισσότερο τις επιτροπές και όχι τις πολιτικές ομάδες, διότι οι δημοσιονομικοί ελεγκτές ε, πίστευαν ότι θα έπρεπε η ΣΕΠΟΛ να μεταφερθεί στην Χάγη και για το θέμα αυτό η καθήλια αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είχε διαφορετική άποψη γιατί στη Χάγη γιατί εκεί ήδη βρισκόνται άλλες δύο, άλλοι δύο οργανισμοί που ασχολούνται με τα θέματα της επόλτη, Eurojust και Europol. Εμείς λοιπόν ε, ελπίζαμε ότι αν όλοι μαζευτούν στην ίδια πόλη, θα υπάρξουν συνέργειες και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει και σημαντική εξοικονόμηση κονδυλίων. Διότι, συνάδελφοι, σημαίνει το εξή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Κυριακή γίνονται προτάσεις ε, για εξοικονόμηση και τη Δευτέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τέλος πάντων, η ΣΕΠΟΛ αντί για τη Χάγη πήγε στη Βουδαπέστη. Ωραία πόλη και η Βουδαπέστη, όμως η άποψή μας σχετικά με την εξοικονόμηση κονδυλίων ε, προφανώς ε, αποδείχθηκε άχρηστη. Τώρα λοιπόν η ΣΕΠΟΛ καλείται να τοποθετηθεί και ε, κατ' ουσίαν, επειδή δεν αλλάζει τίποτα για τις δραστηριότητες της ΣΕΠΟΛ και τίποτα στην εσωτερική της ε, οργάνωση, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού θα είναι πολύ λιτή και εγώ Έχω καταθέσει μόνο λίγες τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο η ΣΕΠΟΛ να συνεργαστεί ή δυνατόν και με άλλες υπηρεσίες και βεβαίως ε, εάν ε, τώρα οι υπόλοιποι οργανισμοί ε, που ασχολούνται με τέτοια θέματα είναι ε, λιγάκι πιο μακριά, κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, παρόλα αυτά πρέπει να συνεργάζονται. Το μόνο έτσι μια εχμή που έβαλα ήταν η εξή. Τη Βουδαπέστη, ε, συγγνώμη κύριε Ντόιτσε, δεν μην το πάρετε προσωπικά, αλλά εγώ τη Βουδαπέστη θέλω να την θεωρούμε ως προσωρινή έδρα της ΕΠΟΛ. Δεν είναι ε, σπόντα για την Ουγγαρία, αλλά είναι μια σπόντα δική μου που διαφωνώ με το να πάει η ΣΕΠΟΛ ε, στη Βουδαπέστη. Άποψη που τη στήριξε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Που και αυτοί βέβαια είχαν τα δικά τους επιχειρήματα που δεν ήταν και αρνητικά ή άσχημα, αλλά μέχρι εγώ είχα διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Να διευκρινίσω. Με συγχωρείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ ότι και απέναντι στην ε, Ουγγαρία θα υπάρχει τέτοια ευγενική στάση, όπως είχα εγώ απέναντί σας, αλλά τέλος πάντων δεν ήθελα να πω αυτό τώρα από δημοσιονομική σκοπιά. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε αυτά που μας παρουσίασε μόλις τώρα και αυτά που υπάρχουν ως μορφή τροπολογίας. Εγώ Συμφωνώ με την προσέγγιση η έδρα των ευρωπαϊκών ε, με την άποψη ότι η έδρα των ευρωπαϊκών οργανισμών ε, δεν ε, την χάνει του κατάλληλου σχεδιασμού. Και δυστυχώς αυτή η έλλειψη σοφροσύνης δεν βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων. Και επίσης, συμφωνώ με την ιδέα ότι ίσως ε, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα αν ε, ομαδοποιούμε οργανισμούς. Πρόκειται για μια προσέγγιση επί της αρχής, για ένα θέμα αρχής. Όμως εδώ δεν ε, μιλάμε για μια οικονομική στρατηγική. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει άλλους στόχους. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν η Ευρωπόλ και η ΣΕΠΟΛ να μην συγχωνευτούν. Μπορεί να μας αρέσει ή να μας αρέσει αυτή η απόφαση. Η ΣΕΠΟΛ έφυγε μόλις από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις βρήκαν μία νέα έδρα και πρόκειται για τη Βουδαπέστη. Εμείς ε, θεωρούμε ότι από δημοσιονομική σκοπιά θα εξοικονομήσουμε πόρους. Η Βουδαπέστη κέρδισε το διαγωνισμό εντός του Συμβουλίου. θέτοντας ε, στη διάθεση της ΕΠΟΛ για 10 χρόνια τις απαραίτητες υποδομές. Αυτές οι υποδομές μόλις εγκαινιάστηκαν στις 6 Νοεμβρίου πριν ένα μήνα και μόλις ε, μετακόμισε η Ακαδημία στη Βουδαπέστη, έτσι λοιπόν κάναμε εξοικονόμηση πόρων. Γιατί, επαναλαμβάνω, εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον για 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να δαπανίσει χρήματα για την Αστυνομική Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, υπό το φως όλων αυτών και από τη δημοσιονομική σκοπιά και από νομική σκοπιά, η τροπολογία αυτή που μόλις κατατέθηκε είναι απαράδεκτη, γιατί ήδη έχει ληφθεί η απόφαση. Όπως και να έχει, η Ευρωπόλ και η ΣΕΠΟΛ έχουν οριστικές έδρες. Αυτή η τροπολογία θέλει να επιφέρει αλλαγές σε αυτό το οριστικό καθεστώς των εδρών. η έδρα στη Βουδαπέστη μας ε, διασφαλίζει ότι θα κάνουμε εξοικονόμηση και εγώ νομίζω ότι είναι και λογικό και σόφρον να υποστηρίξουμε αυτή την έδρα για τις ΕΠΟΛ. Κατά τα λοιπά, εγώ υποστηρίζω να έχουμε ε, ουσιαστικά μια λογική στάση απέναντι στο πώς ε, επιλέγουμε τις έδρες των ευρωπαϊκών οργανισμών, όμως εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόεδρος, εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει και σε άλλη επιτροπή, γιατί στη ΛΥΜΠΕ θα γίνει ακρόση του ηγετή στις 11 Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 16 Δεκεμβρίου και στην Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσουμε είτε στις 19 είτε στις 20 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει το Φεβρουάριο, αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί και ο θέατης στην Ολομέλεια θα γίνει εν καιρό. Τέλη Φεβρουαρίου ή Μάρτιο. Λοιπόν, δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο για αυτό το θέμα, οπότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν για την έκθεση Gerard Depré για τον προϋπολογισμό 2014 τμήμα 3 και μεταφορές μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας τάση. Καταρχήν θέλω να μιλήσω για τη μεταφορά 42 και θα ήθελα να σας εκκοινώσω ένα διπλό καλό νέο. Καταρχήν, η κυρία Γκρέσλε έχει υποβάλει κάποιες αντιρρήσεις και ήθελε πρόσθετες ε, πληροφορίες από την Κομισιόν, τι έλαβε, είναι ικανοποιημένη λοιπόν και αυτό θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε σήμερα. Δύο. Για το περιεχόμενο, για το τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω δύο στοιχεία τη νέα σελίδα της Κομισιόν. Είναι, μια είναι ένα νέο μεγάλο. Δεν θα αντικατοπτρίζει πλέον μόνο το εσωτερικό οργανόγραμμα, αλλά θα επικεντρωθεί πραγματικά και στις ανάγκες και στις προσδοκίες των χρηστών. Αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο. Έτσι λοιπόν τώρα εκπονείται και μια πολιτική για τη χρήση των γλωσσών και θα μπορεί η Κομισιόν να απευθύνεται στους πολίτες τη μητρική τους γλώσσα. Αυτό είναι λοιπόν το διτό καλό νέο που είχα να σας ανακοινώσω για αυτή τη μεταφορά υπαριθμό 42. Ευχαριστούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον υπαριθμό 37 μεταφορά, πρόκειται για μια σημαντική μεταφορά των 44 εκατομμυρίων 200.000 ευρώ θα κάνουμε πραγματικές οικονομίες ό,τι αφορά τι διοικητικέ γραμμές των εκτελεστικών οργανισμών που θα πάνε προ τι επιχειρησιακέ γραμμές του προγράμματος Ορίζοντα 2020, πολιτική μεταφορών, ΣΥΝ και αυτό μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα εσωτερικής ανακατανομής του προϋπολογισμού ε, σημαντικό ποσό. Σε ό,τι αφορά τώρα την τρίτη μεταφορά, υπαριθμών 53 πρόκειται για 1,25 εκατομμύρια από την οποία των προγραμμάτων της περίοδου 2000-2006 που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε εκαθάριση τεκρεμών λογαριασμών υπέρ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Γεωργικού Ταμείου Εγγύησεων. Και θα ήθελα να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι με αυτές τις τρεις μεταφορές. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις υπάρχουν. Διαφωνείτε να ψηφίσουμε συνολικά και αυτές τις τρεις μεταφορές. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Έτσι λοιπόν ε, όσοι εγκρίνουν αυτές τις τρεις μεταφορές να το δηλώσουν με ανάταση χειρός παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Δεν βλέπω να υπάρχουν αρνητικές ψηφί. Αποχές ούτε. Δύο αποχές. Λοιπόν, αυτές οι μεταφορές εγκρίνονται. Ελπίζω ότι το ίδιο θα ισχύει και για το Συμβούλιο, ότι θα υπάρχει έγκριση. Κυρία Χολμάιερ, για τα υπόλοιπα τμήματα, προπολογισμό 2014 και πάλι εδώ έχουμε κάποιε μεταφορέ. Έχουμε και το 55, λέει ο κύριος Δεπρέ. Απλώς να παρουσιάσω το 55, αλλά κυρία Χολμάιερ. Όχι, όχι για το 55, γιατί αφορά την πολιτική για τα κτίρια. Μπορούμε να ζητήσουμε την κυρία Χολμαέρ να το παρουσιάσει γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο Λουξεμβούργο στο κτίριο Ζαν Μονέ όπου βρήκαμε αμίαντο και είναι επικίνδυνο για όλους όσους ε, εργάζονται σε αυτό το κτίριο αλλά νομίζω ότι θα τα πείτε καλύτερα από μένα παρακαλώ. Μάλιστα θα φτάσουμε και σε αυτό όταν συζητήσουμε για τα κτίρια. Πολιτική για τα κίνητα. Παρακαλώ, κυρία Χολμάιερ. Λοιπόν, το θέμα των ε, κτηρίων, εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας στείλει τα διάφορα στοιχεία. Πρόκειται για το κτίριο Ζαν Μονέ, το οποίο δυστυχώς ε, κρίνεται επικίνδυνο λόγω του αμοιάντου για όσους ε, εργάζονται στο κτίριο αυτό. Άρα δηλαδή θα πρέπει να δαπανίσουμε πολλά κονδύλια έτσι ώστε να βρούμε κάποια άλλη προσωρινή ε, στέγαση για τους ε, συνεργάτες μέχρι να επισκευάσουμε τον Ζαν Μονέ. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε εκεί τους ε, συνεργάτες γιατί θα είναι εκτεθειμένοι σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Τις απαραίτητες πληροφορίες θα τις πάρουμε σύντομα και τότε θα μπορούμε να οργανώσουμε και τη μεταφορά. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, ακόμα και αν είναι ακριβό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στο κτίριο αυτό τους συνεργάτες μας, το προσωπικό Παλαιότερα, από ό,τι φαίνεται, τα κτίρια κατασκευάζονταν ε, χωρίς ε, καμία μέρημνα για τον αμύοντο, ο οποίος ε, βρίσκεται μέσα στους τοίχους. Είναι αδύνατον αυτό να παραμείνουν εκεί οι άνθρωποι για τρία χρόνια. Δεν μας αρέσει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ε, θα πρέπει να εκταμιεύσουμε πολλά κονδύλια κύριε Πρόεδρε. Και αν όμως το συγκρίνεται αυτό σε σχέση με τα ποσά τα οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη, θα τρομάξετε. Τέλος πάντων δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι. Και πάω τώρα, κύριε Πρόεδρε, έχω πολλά να πω. Τα ε, κάνω σύντομα. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 55.000 ε, ευρώ θέλει για να ε, κάνει κάποιες βελτιώσεις στη μηχανογράφηση. Αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εξοικονόμησε αυτό χρήματα σε ε, θέματα ενέργειας. Θέλετε να τα πω σε ομάδες, πώς θέλετε να τα πω. Κύριε Πρόεδρε, πώς όλα μαζί. Λοιπόν, Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία επιθυμεί να αυξήσει τον προπολογισμό του για ταξίδια και αυτό να το αφαιρέσει από μια άλλη γραμμή του προπολογισμού της τάξης των 50.000 και αυτό γίνεται. Το δεύτερο που θέλουν είναι να αυξήσουν ε, κατά 45.000 τον τεχνικό του εξοπλισμό των fitting out of premises, δηλαδή ε, θέλουν να βελτιώσουν το σύστημα θέρμανσης, ε, να περάσουν στο αέριο για να είναι έτσι πιο φιλική προς το περιβάλλον και με μικρότερο κόστος, πάλι 45.000 ευρώ. Και επιπλέον επιθυμούν βελτίωση του μηχανογραφικού τους και πάλι ε, σε θέματα λογισμικού <clears throat> και διατήρηση του εξοπλισμού τους. 148.680 ευρώ. Εδώ εντάσσεται και η πύλη για τα μέλη, έτσι ώστε τα μέλη της Επιτροπής ε, να μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα την πύλη αυτή. Κατόπιν ε, ο μάνατζερ του intranet και του extranet και επίσης να μην διατίθενται έγγραφα αλλά περισσότερο ε, μέσω του διαδικτύου 748.680 ευρώ. Επίσης θέλουν τεχνική εγκατάσταση να τη βελτιώσουν σε άλλους τομείς και εδώ χρειάζονται άλλες 27.000 και 420 ευρώ. Και το τελευταίο που αφορά στην Επιτροπή των Περιφερειών είναι αυτό. Χρειάζονται 925.000. Αυτό προκύπτει από τιμαριθμική προσαρμογή των μισθών του προσωπικού που όμως καταπίπτει και μέσω αυτό το ποσό θέλουν να το καταβάλουν για τα leasing έτσι ώστε του χρόνου να έχουν κάποιες διευκολύνσεις σε θέματα τη μαριθμική αναπροσαρμογής και οτιδήποτε άλλο παρεμφερές. Θέλουν λοιπόν φέτος να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 925.000 για να μπορούν να τις μεταφέρουν επειδή έχουν περισσέψει και κατόπιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κονδύλι είχαμε αποφασίσει το κτίριο ΚΑΝΤ να μην συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αλλά το ραμασάζ να μαζέψουμε όλα τα υπόλοιπα που προκύπτουν για να πληρώσουμε του χρόνου τους λογαριασμούς. Μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στα 71 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή θα μεταφέρουμε 71 εκατομμύρια. Και είχαμε τύχη στις μεταβατικές δαπάνες. Οι δαπάνες για τους βοηθούς είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε προβλεφτεί αρχικά. Εξοικονομήσαμε δαπάνες και στα μέλη 38 εκατομμύρια προέρχονται από τον τομέα των μεταβατικών δαπανών που δεν μπορέσαμε να εκταμιεύσουμε. Τα υπόλοιπα προέρχονται από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγκαστούμε να αναλάβουμε χρέη, να αναλάβουμε, να ζητήσουμε δάνεια. Το βρίσκω πάρα πολύ θετικό αυτό, το να μην είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε σε δανεισμό για το κτίριο CAD και είχαμε συμφωνήσει ότι θα ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο. Επίσης έχουμε μετά την ε, ΟΚΕ που και αυτοί επιθυμούν να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους, το μηχανογραφικό τους. Ε, μιλάμε για 989.000 ευρώ και τελευταίος είναι ο Ombudsman, ο διαμεσολαβητής, που ζητάει μεταφορά 155.000 ευρώ. Αυτές τις 155.000, μισό λεπτό να το δω κι εγώ, προέρχονται από τη μετάφραση και τη δημοσίευση για να καλύψει ανάγκες σε, σε θέματα μισθοδοσίας, λόγω ε, τιμαριθμικής προσαρμογής της τάξης του 0,8%. Αυτά θέλουν να εγγράψουν στον προεπλογισμό τους και θα το επιτύχουν με αυτή τη μεταφορά κονδυλίων που σας ανέφερα. Προσπάθησα να είμαι σύντομη. Η συντομία, σαφήνεια και ταχύτητα, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια για όλα αυτά. Κύριε Βέστρε. το Κυρία Κρέσλε, λοιπόν, ε, εκπλήσωμε λιγάκι ως προς το ότι ε, παραμένουν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ε, στους βοηθούς των βουλευτών. Εμάς μας είχαν πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ χρειάζομαι συνεργάτες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι δεν το βρίσκω καλό αυτή την πληροφορία να την έχετε γράψει κάτω-κάτω και στο τέλος του όλου εγγράφου να πρέπει κανείς να ψάξει να... Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση. Κοιτάξτε, ε, αυτή η γραμμή δεν θα υπάρχει το 2015. Είχαμε σκεφτεί ότι αν προκύψουν επιπρόσθετες δαπάνε για αποχωρώντα μέλη και αποχωρώντες βοηθούς, θα ε, χρησιμοποιούσαμε αυτά τα κονδύλια αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το 98% των βοηθών θα επαναπροσλαμβάνονταν, μπορούσε να, θα μπορούσε να είναι 40% ή 50%. Ε, εμείς ε, το είχαμε σκεφτεί διαφορετικά και τώρα πια το 15 όλα αυτά δεν θα προβλέπονται. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν στο κτίριο αυτό, τι απομένει να πληρωθεί παρακαλώ. Τι χρειάζεται ακόμα να πληρωθεί για αυτό το κτίριο μετά ε, το έμβασμα, τι θα χρειαστεί ακόμα για να έχω καθαρή καρδιά. Νομίζω ότι είναι σφάλμα να μην ε, κάνουμε τις εκτιμήσεις τον προπολογισμό για να έχουμε σαφήνεια. Τελικά, κάνουμε αυτό που έκανε και το Συμβούλιο με το Residence Palace. Και είναι σφάλμα, διότι δεν μπορούμε έτσι να κατακρίνουμε τους άλλους όταν κάνουμε και εμείς τα ίδια, όταν τους λέμε ότι δεν μας λένε ακριβώς τι χρειάζονται. Monsieur Arnott. yes, I'm just wondering um, the first... Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ε. Το πρώτο το οποίο συζήτηθη ήταν ε, η ασφάλεια και η υγεία. Αφορά τον αμίαντο. Και νομίζω αν θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό πραγματικά. Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab. Για τον Jean Monnet μιλάμε. Bon. Retirez votre demande de vote séparé. Madame. Αποσύρετε λοιπόν το έτοιμά σα για ξεχωριστή ψηφοφορία. Τι απομένει τώρα εδώ πέρα για, για πληρωμή. Αυτή τη, στιγμή, ναι. αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Χρειαζόμαστε ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη περικοπή στις δαπάνες. Σεβόμαστε πλήρως ε, τα δημοσιονομικά σχέδια που έχουν συμφωνηθεί από την ε, Δημοσιονομική Επιτροπή μετά την επισκέψη της στο Λουξεμβούργο και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και λάθη. Στον προπολογισμό μας ε, δεν έχουμε λάθη, ούτε καν για 1%. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι είχαμε ε, μία χρονιά εκλογική με πάρα πολλές ε, αβεβαιότητες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Εκτελούμε πάρα πολύ καλά τον προϋπολογισμό μας. Και διαθέσιμα ποσά θα τα χρησιμοποιούσαμε για να μην ζητήσουμε περαιτέρω πιστώσεις. Την επόμενη φορά θα σας φέρω το πλαίσιο γιατί έτσι θα μπορείτε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Θα τα θέσω όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Την επόμενη χρονιά πρέπει να προβλέψουμε να πληρώσουμε 85 δισεκατομμύρια, ενώ τώρα πληρώνουμε 75. Φτάνουμε σε μια χρηματοδότηση 86 εκατομμυρίων που 186 εκατομμυρίων που αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού κόστους. κόστους. σιγά σιγά στο 50% της χρηματοδότησης του έργου. Λοιπόν, από πλευράς όμως σαφήνειας, ε, δημοσιονομικής σαφήνειας, ε, δεν θα ήταν καλό να εγγράφονται τέτοιες διαδικασίες στον προπολογισμό. Τέτοια έργα, μεγάλα έργα, αν κατάλαβα καλά, οι επιστώσεις γράφηκαν με μεταφορές, αλλά αυτά τα 71 εκατομμύρια τελικά, με συγχωρείτε, κάνει κρύο σε αυτή την αίθουσα, κρυώνουμε. Οικονομία στη θέρμανση κάνουμε, τι γίνεται. Χρειάστηκε να φορέσω το κασκόλ μου γιατί κρυώνω. Bon, euh, fait des économies pour financer l'immeuble Conrad Adenauer οικονομίες για να μεταδοτήσουμε το, κτίριο Conrad Adenauer. Bon, je pense que les membres de la commission sont suffisamment éclairés. Νομίζω ότι έχουμε πλέον αρκετές πληροφορίες για να ψηφίσουμε. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε όλα τα όσα προτείνει η κυρία Ολμέγερ. Όχι. Ποιοι είναι υπέρ, ψηφίζουμε τώρα, ποιοι είναι υπέρ της έγκρισης των μεταφορών που προτείνει η κυρία Ολμέγερ να σηκώσουν το χέρι. Ευχαριστώ. Κατά. Όχι. Κάποιος δεν συμφωνεί. Ένας μόνον. Αποχές. Τρεις αποχές. Συνεπώς ε, είναι θετική η έκβαση της ψηφοφορίας. Nous avons maintenant euh, dans la politique euh, immobilière création. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη δημιουργία ενός ε, χώρου υποδοχής επισκεπτών στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Κυρία Χολμάιερ. Es geht hier heute um eine grundsätzliche Zustimmung. Wir haben Πρόκειται για μια συμφωνία επί της αρχής. Ε, το 2014 έχουμε 2,5 ε, εκατομμύρια κόστος και επί της αρχής ελήφθη απόφαση. Δύο φορές αυτή την Επιτροπή έχει υπάρξει έγκριση, αλλά πάρα πολλοί μας ρωτούν γιατί όλο αυτό το θέμα θεωρείται εμπιστευτικό. Γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες και δεν ξέραμε πώς θα το καλύψουμε οικονομικά. Πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι λοιπόν, Εμείς ε, στηριχτήκαμε στην γραμματεία για να δώσει ενημέρωση στους συναδέλφους ε, σήμερα για να έχουμε ένα νέο κέντρο επισκεπτών ε, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα λεωφορεία που καταφτάνουν εδώ και ξέρετε, οι άνθρωποι κινδυνεύουν γιατί κατεβαίνουν από το λεωφορείο μέσα στη μέση του δρόμου που υπάρχει κίνηση. Και ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το σχεδιασμό προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει μια διαφορετική υποδοχή των επισκεπτών κατά την άφηξή τους εδώ στα κτηριά μας. Έχουμε ε, μια επιφάνεια 320 τετραγωνικών ε, και θα υπάρχουν και τουαλέτες 110 τετραγωνικά και ένας χώρος όπου θα μπορούν να κάθονται οι επισκέπτες. Όλοι γνωρίζουν ε, πόσα πολλά λεωφορεία έρχονται και μερικές φορές οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ουρά μπροστά από την ε, πόρτα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, επειδή παίρνουν και αυτοκίνητα, πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Ήδη δύο φορές έχουμε επιβεβαιώσει το ποσό και δεν θα αλλάξει αυτό. Και Κατόπιν θα έχουμε και ακόμα 170 τετραγωνικά άλλους χώρους που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για να στεγάσουμε τεχνικές υποδομές. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παροβιλαντικές πτυχές και θα πρέπει να οργανώσουμε διαφορετικά και το θέμα της ασφάλειας. Σήμερα καθυστερούν πάρα πολλοί επισκέπτες για να περάσουν τον έλεγχο Νομίζω ότι θα πρέπει να το επιταχύνουμε αυτό. Δεν θέλουμε να είναι πολύπλοκα τα πράγματα για το κοινό. Θα υπάρχει και μια επίσημη διαδικασία διαγωνισμού. Αποφασίσαμε ότι όλο το κόστος θα είναι 2,5 εκατομμύρια. Και για του χρόνου 2,656 και για τον επόμενο 2,44 εκατομμύρια. Όλα αυτά για να έχουμε ένα κατάλληλο χώρο υποδοχής για τους επισκέπτες και να κάνουμε τις διάφορες προσαρμογές στον εφιστάμενο χώρο επισκεπτών για όσους παρευρίσκονται και σε συνεδριάσεις. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει στο κτίριο PHS, το οποίο παλιώνει και αρχίζουμε να βλέπουμε ήδη κάποια προβλήματα. Ξέρετε, αυτό θέλουμε να το κάνουμε ε, καταρχήν και κατόπιν να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσετε για αυτό το ποσό για το 2,656 και το 2,44 για του χρόνου. Εάν έχετε ερωτήσεις, δεν ξέρω αν υπήρξαν άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ, όποιος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε η κυρία Χολμάερ ηχούν ε, λογικά, ε, δηλαδή επί του περιεχομένου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά ξέρετε, εγώ ζήτησα το λόγο ως ε, νέα βουλευτής και ως σκιώδης εισηγήτρια, γιατί θέλω να σας πω ότι με εκπλήσει λιγάκι ε, το θέμα της ε, πληροφόρησης. Ε, εδώ πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη απόφαση, γιατί πρόκειται για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Και κατά την άποψή μου, τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει καταρχήν να υποβάλλονται στις πολιτικές ομάδες και να ελέγχονται. Θεωρώ λοιπόν ότι άλλες πολιτικές ομάδες δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Εγώ τα ζήτησα χθες ε, και μου έδωσαν ε, και μία εισήγηση σε PowerPoint ε, που δεν μπορεί όμως να ψηφιοποιηθεί κατόπιν τούτου δεν μπορούσε κανείς να κάνει και πολλά πράγματα με αυτή την παρουσίαση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει κανείς να έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να ξανασυζητήσει από αυτών των θεμάτων.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 πρέπει να τα αναβάλουμε για την επόμενη φορά. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους ε, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις, άρα είμαστε κάτω από πίεση χρόνου. Και υπάρχει και ένα λάθος που έχει γίνει μέχρι τώρα. Κανείς δεν μου είπε ότι υπάρχει κάποιος σκιώδη συγητής. Και μέχρι τώρα η ήταν ότι τα έγγραφα ε, δίδονται απόρριτα ανάμεσα στους ε, σκιώδης ηγητές. Και όταν κάποιος ε, πει ότι είναι σκιώδης ηγητής, τότε παίρνει αυτά τα απόρριτα έγγραφα. Γιατί ξέρετε, είναι απόρριτες οι πληροφορίες, γιατί αν τις δημοσιοποιήσουμε, τότε ενδέχεται να προβούμε σε παρανομίες και παρατυπίες. Γι' αυτό δεν δίνουμε όλα τα έγγραφα στο σύνολό τους. Τα δίνουμε μόνο, επειδή είναι απόρριτα, στους ε, εισηγητές και οδησηγητές και στους συμβούλους. Βεβαίως, ε, τα ποσά επιβεβαιώθηκαν δύο φορές. Δεν θα αλλάξουν τα ποσά, ούτε θα αυξηθούν, ούτε θα μειωθούν. Έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό. Αυτό έχει γίνει σε αντίθεση με το κτίριο ΚΑΝΤ και ενεγράφησαν ήδη την προηγούμενη φορά. Μόνο που εσείς επειδή είστε νέα, γι' αυτό δεν ενημερωθήκατε. Δεν ενημερωθήκατε ότι αυτά έχουν εγγραφεί στον προπολισμό. Τα ποσά δεν θα ξεπεραστούν, δεν θα αλλάξει τίποτα στα ποσά, θα παραμείνουμε μέσα στον προπολογισμό, μόνο που ολοκληρώνει κανείς τον προγραμματισμό, τον οποίο, επί του οποίου έχουν ήδη ληφθεί δύο φορές αποφάσεις. Δεν μπορούμε εδώ να μιλήσουμε δημόσια για τις λεπτομέρειες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατηδίαν, ε, διότι αλλιώς ε, θα θέσουμε σε κίνδυνο τον προγραμματισμό που δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη γιατί μέχρι τώρα ε, δεν μου είχε πει κανεί ότι υπάρχει σκιώδη εισηγητή. Δεν υπήρχε σκιώδη συγητή. Ε, τώρα μου το είπατε και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχω και σκιώδη εισηγήτρια. Και χαίρομαι που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κατηδίαν. Βεβαίω ε, πρέπει να σα πω ότι να ξέρετε είμαστε υποποίηση χρόνου. Δεν θα υπάρξει τίποτα το καινούριο, έχουν εγγραφεί τα ποσά στον προπολογισμό, αυτά που έχουμε αποφασίσει ήδη δύο φορές, μόνο που τώρα πρέπει να λάβουμε την τελική και αμετάκλητη απόφαση. κυρία Κρέσλε, έχω ε, μία ερώτηση. Αν όλα είναι ξεκάθαρα, τι να αποφασίσουμε. Και τι να αποφασίσω εγώ, κάτι που δεν ξέρω τι, ποιο είναι το περιεχόμενό του. Εκλεγμένη βουλευτή είμαι. Ε, πού το λέτε εσείς τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Εμένα με έχουν εκλέξει βουλευτή και δεν μου είπανε θα είσαι εισηγήτρια ή σκιώδη ή παρεμφερή. Βουλευτή μου είπανε ότι θα, βουλευτής θα είμαι. Κοιτάξτε, έχουν διανεμηθεί τα στοιχεία σε όλα τα μέλη, λέει η κυρία Χολμάιρα. Κοιτάξτε, τώρα, Ακόμα και αν έγινε αυτό το λάθος με τη, το σκιόντι σιγήτρα ή όχι, δεν το ξέρω τι έγινε, αλλά εγώ ε, θέλω λιγάκι να το δω το θέμα, να, το διαβάσω, το μελετήσω. Τώρα δεν μπορώ να ευλογήσω κάτι που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν το γνωρίζω το θέμα. Σας παρακαλώ για την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη συνεδρίαση να ψηφίσουμε. Κυρία η κυρία Χολμέγερ μα είπε ότι έπρεπε να πάρουμε μια θέση πριν από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αν το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ίσως ε, η απέναντι Γενική Διεύθυνση μπορούν να μας πούνε ε, σχετικά με την πίεση χρόνου να μας ενημερώσουν για να ξέρουμε και εμείς τι θα αποφασίσουμε. Κυρία Κρέσλε, μισό λεπτό. Ε, εγώ το είδα αυτό το έγγραφο, αλλά δεν μπορώ από το έγγραφο να καταλάβω ότι είναι υποβλήθηκε η απόφαση, θα ήταν καλό να μας εξηγήσετε λιγάκι, να μας δώσετε και κάτι άλλο να καταλαβαίνουμε. Εγώ δεν είδα καμία PowerPoint, εισήγηση με PowerPoint. Ε, Ευχαριστώ μισό λεπτό. Α, θα μου άρεσε να δω κάτι, λέει η κυρία Κρέσλε. Λοιπόν, ο κύριος Κλετή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, θα μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ μια διευκρίνηση για αυτό το θέμα του απορρίτου. Νομίζω ότι απλώς ε, εδώ ε, θίξαμε ακροθυγός το χρηματοκονισμό που προβλέπει στο άρθρο 203 παράγραφος 5 ε, ότι τα έγγραφα που κοινοποιούνται σε σχέση με τα κίνητα είναι εμπιστευτικά. Προφανώς όλος ο φάκελος διαβιβάστηκε στο πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών και νομίζω ότι ήταν στη διάθεσή σας στο πλαίσιο εμπιστευτικής συζήτησης προκειμένου ο κάθε βουλευτής να μπορέσει να γνωρίσει όλα τα στοιχεία χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό ήταν ένα μέτρο προστασίας προκειμένου αυτές οι πληροφορίες να μην αποκαλυφθούν στο διαδίκτυο κτλ γιατί κάτι τέτοιο θα μας έβαζε σε δύσκολη θέση, καθώς τρέχει η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τώρα το ίδιο το project συζητήθηκε κατά την υιοθέτηση του ε, προσωρινού προπολογισμού, γιατί είχαμε εγγράψει στον προπολογισμό ένα ποσό, στον προπολογισμό του 2015, και για να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε, υπάρχουν δύο επίπεδα προσφυγής ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού, μια προκαταρκτική διαδικασία, διαδικασία, άρθρο 203, εδάφιο 3 και είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο όπου όταν υπάρχουν προσφορές επιτάπητος μπορούμε να πούμε ότι πράγματι το συνολικό κόστος θα ήταν 5.200.000 για ένα έργο που είχε θετηθεί και από το Προεδρείο και από την Επιτροπή του Προπολογισμού στο στάδιο της έσχατης παρουσίασης. Ίσως ε, είναι κάπως πολύπλοκο το σύνολο και θα πρέπει ίσως να γνωρίσουμε ότι καθώς αλλάξαμε και θητεία θα πρέπει να επενθυμίσουμε κάποια στοιχεία αλλά εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε ε, πραγματικά σε μια διαδικασία η οποία δεν ε, έχει διακοπή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ακούστε, καθώς Μπορούμε αυτό το θέμα να το δούμε στις 11 του μήνα, καθώς έχουμε πάλι συνεδρία της Επιτροπή μας. Θα πρότεινα τότε να ψηφίσουμε. Παρακαλώ, κύριε Κρέσλε. Κοιτάξτε, εγώ απλώ είπα ότι αν είναι διαθέσιμα τα έγγραφα, δεν ε, μου είπε κανεί ότι αν μπορεί να πα εκεί να δει αυτά τα έγγραφα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω τώρα να δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά αρνούμε να ψηφίσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα δαπανίσουμε εδώ όλη τη βραδιά. Την επόμενη βδομάδα προτείνω να ψηφίσουμε και έτσι να έχετε και χρόνο να δείτε και τα έγγραφα. Κυρία Χολμέγερ. Προς ενημέρωσή σας, οι βασικές πληροφορίες για το project αυτό μπορούν να διατεθούν, υπάρχουν για όλα τα μέλη με τη μορφή PowerPoint, ήδη και σήμερα. Πρόκειται μόνο για τα στοιχεία, για τις εταιρείες. Αυτό δεν το δημοσιοποιούμε και συνειδητά μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία, υπάρχει λόγος κοινοποιούνται μόνο ε, στους εισηγητές και επ' αυτού έχουμε συμφωνήσει η Επιτροπή. Κατά τα άλλα όλοι μπορούν να δουν τι είναι το κτίριο, πώς προγραμματίζεται, τι μορφή θα λάβει. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο PowerPoint. Ε, επ' αυτού δεν υπάρχει τίποτα το απόρριτο. Μόνο που δεν σας βάλαμε μπροστά σας την ε, παρουσίαση PowerPoint ε, και με μορφή χαρτιού. Σας δώσαμε τη δυνατότητα να ψάξετε στο διαδίκτυο γιατί εκεί εκεί μπορείτε να τα δείτε και καλύτερα. Είναι πιο καθαρές οι φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, όταν θα το έχετε δει, θα τοποθετηθούμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, είπα τα διάφορα, κάποια θέματα. Όχι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ολοκληρώνω τη συνεδρίαση.